ώστε και εμπράκτος αυτέ τι συστάσεις. Γιατί θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά του και να έχουν αξιοπρέπεια και ισότητα. Σα ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, κύριε Ματίας, ευχαριστώ όσου έλαβαν μέρο στη συζήτηση. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε, θα ψηφίσουμε αύριο από τι 12. Ήδη έχουμε σχεδόν ημίωρη καθυστέρηση σε σχέση με το επόμενο θέμα. Θα προσπαθήσουμε να βιαστούμε όσο γίνεται. Η πρώτη ερώτηση είναι η ερώτηση 14 σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών πιστώσεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων του κυρίου Νικουλέσκου. Όταν είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να δώσει την απάντησή της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συμφωνεί με την ερώτηση αυτή και το άρθρο στην εφημερίδα Financial Times, γιατί έτσι θα συμβάλλουμε στην ε, αποτελεσματικότητα των διαρθρωτικών πολιτικών και ιδιαίτερα της συνοχής. Ήδη έχουμε μία αργή ανάκαμψη και τα πιο ενημερωμένα στοιχεία δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πραγματοποίησε στο πρώτο εξάμεινο του 2010 πολύ περισσότερες ε, πληρωμές από ό,τι στο παρελθόν. Οι περισσότερες πληρωμές ήταν ενδιάμεσες πληρωμές ήταν επιστροφές ταπανών που είχαν γίνει και επιστοποιηθεί στα κράτη-μέλη. Και έτσι είχε γίνει και στι προηγούμενες περιόδους, αλλά φαίνεται ότι επιταχύνεται ο ρυθμός πληρωμών και μάλιστα η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων από τα κράτη-μέλη είναι στο 21% για το Ταμείο Συνοχής, 22% για το Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξη και 23% για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σε ό,τι αφορά την ε, υποστήριξη για πολυεθνικές και μεγάλες εταιρείες, ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο βασικός στόχος της ε, πολιτικής συνοχής είναι η οικονομική μεγέθυνση και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για συγκεκριμένες περιοχές και κράτη-μέλη. Οποιαδήποτε υποστήριξη των παραγωγικών επενδύσεων θα πρέπει να ειδωθεί από αυτή τη σκοπιά την προώθηση της απασχόλησης και την οικονομική μεγέθυνση. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί είτε με τη σύσταση δίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων είτε με την υποστήριξη μεγαλύτερων εταιριών. Πάντως οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα προγράμματά της ε, στρέφονται κυρίως προς την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως φαίνεται και τα καταστατικά των Ταμείων ε, Κοινωνικού και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είχαμε και, την, ε, και τις διαπραγματεύσεις στα, στα έγγραφα προγραμματισμού και όλα αυτά δείχνουν ότι οι παραγωγικές επενδύσεις ε, στόχο έχουν την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μπορεί βέβαια να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε σε, μικρομεσα... σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αρκεί αυτές να πληρούν τη... τους στόχους των διαρθρωτικών ταμείων ή των σχετικών προγραμμάτων. 57 ε, δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε δώσει μεταξύ του 2007 και 2013 για υποστήριξη επιχειρήσεων και το μεγαλύτερο μερίδιο αφορά την καινοτομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι πολυεθνικές δεν είναι δικαιούχοι της υποστήριξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινωνικού Ταμείου κυρίω. παρόλο που μερικές φορές ε, λαμβάνουν κάποια συγχρηματοδότηση. Το Κοινωνικό Ταμείο υποστηρίζει τους ανθρώπινους πόρους, βελτιώνει τα προσόντα τους και δίνει έμφαση στην κατάρτιση και την επιμόρφωση. Για να μπορεί κάποιος να βρει δουλειά σε μια άλλη εταιρεία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για να παραμείνουν οι εργαζομένοι στην αγορά εργασίας. Δεν μας ενδιαφέρει για την κατάρτιση ε, ούτε το μέγεθος ούτε το όνομα της εταιρείας που παρέχει αυτή την κατάρτιση. Σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να βοηθούμε εταιρείε που περιορίζουν το εργατικό τους δυναμικό. Γιατί έτσι το αποτέλεσμα των επενδύσεων θα είναι μηδενικό, για να μην πω και αρνητικό. Όταν μια εταιρεία κλείνει μέσα σε πέντε χρόνια από την υποστήριξη, τα κονδύλια που έχει λάβει πρέπει να επιστραφούν. Επίσης, το τελευταίο σημείο που είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις που θα πρέπει να γίνουν, αλλά δεν μπορούμε να γνωρούμε τον γενικό στατικό αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εθελοτυφλεί ούτε παραμερίζει τα προβλήματα. Θα συνεχίσουμε τις αλλαγές και τις βελτιώσεις της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική συνοχής ευνοεί τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες ε, περιοχές της Ένωσης, αλλά σίγουρα έχει θετικά αποτελέσματα και για την ε, γενικότερη ευρωπαϊκή επικράτεια. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Νικολέσκου, μετά στον κύριο Ρούμπιχ και μετά στην κυρία Πρινκεβιτσούτε. Ο κύριος Νικολέσκου για τη συμπληρωματική. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την ποιότητα της απάντησης του και των πληροφοριών που μας έδωσε. Αλλά και στη συζήτηση όταν συζητούμε για αυτά τα θέματα θα πρέπει να ασχολούμαστε και με τα μελλοντικά μέτρα για να αποφεύγουμε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Και αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν αυτά τα αποτελέσματα, αν τα μάθει ο κόσμος, μήπως ε, κλονίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Ρούμπεχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως για την ενημέρωση, γιατί αποτελεί τη βάση για μια λογική συζήτηση και τη σαφή ε, προσήλωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί ε, απασχολούν τα δύο τρίτα των ε, εργαζομένων στην Ευρώπη και πληρώνουν το 80% των φόρων οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ερωτώ, στο μέλλον η υποδομή για την έρευνα και ε, τα προγράμματα ε, πλαίσιο δεν μπορούν να ενισχυθούν λίγο περισσότερο ακριβώς σε αυτό το τομέα. Και η κυρία Πλίνκεβιτσιούτε. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε για την απάντηση. Εγώ έχω την εξής ερώτηση. Τα διορθωτικά ταμεία, κυρίως το κοινωνικό ταμείο, έχουν στόχο τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης και τη μετεκπαίδευση των εργαζομένων για να αυξήσουν τα προσόντα και τις δεξιότητές τους. Διεθνώς όμως οι μεγάλες επιχειρήσεις θεωρείται ότι είναι στην ίδια μοίρα με τις μικρομεσαίες. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ σκληρός για την επιδότηση από τα διορθωτικά ταμεία. Εσείς τι πιστεύετε δεν θα μπορούσατε να κάνετε κάποιες προτάσεις διαφορετικές για μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις ε, ή να υπάρχουν οι ίδιοι όροι παιχνιδιού και για τις δύο. Ο Επίτροπος, παρακαλώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Καταρχάς, για την υποδομή, την ερευνητική, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καινοτομία, ήδη από σήμερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και μάλιστα γενναία σε τάξη ε, διψήφια δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της ε, καινοτομίας στην προγραμματική περίοδο 2000-2006, εάν δεν απατώμε, ε, πάνω από 30.000 επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν σε αυτό τον τομέα πάρα πολύ ε, στοχευμένα και επίσης θεωρούμε ότι οι ερευνητικές υποδομές ε, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικές και στο μέλλον. Και πέρα από τον αμυγός οικονομικό τομέα και στην ε, θεμελιώδη έρευνα και αν δυνατόν στην τρέχουσα ακόμα προγραμματική περίοδο θα προτείνουμε ένα πρόγραμμα και στο ΕΣΦΡΙ, στον οδικό χάρτη, για πρώτη φορά αναφέρεται και πρικοδοτείται από τα αντίστοιχα κονδύλια. Διότι απεδείχθη ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα πάρα πολύ αηφόρο και βιώσιμο σε μια περιφέρεια το οποίο εμβέλει επερβαίνει κατά πολύ τη στενή ε, έννοια της εταιρεία και δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης και ε, στους προμηθευτές, όχι στην ίδια την εταιρεία. Γιατί χρειάζεται η θεμελιώδης έρευνα και υποδομές και σέρβις και σε ένα τέτοιο πρόγραμμα στην Ουγγαρία. Για την επόμενη λοιπόν προγραμματική περίοδο θα στραφούμε και προς τα πανεπιστήμια που ε, τελικά θα έχουν ε, συγκεκριμένες επιπτώσεις. Γιατί ήδη από σήμερα στα πανεπιστήμια η έρευνα είναι κατά ένα τρίτο εφαρμοσμένη έρευνα που είναι υπέρ της ε, οικονομίας και δημιουργεί βιώσιμες θέσεις απασχόλησης. Σε ό,τι αφορά τα όσα ρώτησε η κυρία συνάδελφος, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Κατά κανόνα, οι εργαζόμενοι ή οι άνεργοι ε, ενισχύονται με μετακπαίδευση, με κατάρτιση έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιούν και να βελτιώνουν τις δυνατότητες που έχουν για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Είτε αυτό είναι στο εσωτερικό της ίδιας εταιρείας στην οποία εργάζονται, είτε στην περίπτωση των ανέργων για να αυξήσουν τα προσόντα τους και τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν ε, το προφίλ τους για να μπορέσουν να ε, απασχοληθούν σε κάποια άλλη θέση εργασίας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ίσως αυτό να εννοείτε, Γιατί πάντα επικρίνεται το γεγονός ότι για τους υπαλλήλους της McDonald's ε, προτάθηκαν σεμινάρια μετεκπαίδευσης. Θα πρέπει να γίνει μια διάκριση εδώ όμως. Ήταν μετεκπαίδευση και κατάρτιση για υπαλλήλους του McDonald's για να μπορούν στη συνέχεια να έχουν περισσότερα προσόντα για την αγορά εργασίας. Γνωρίζετε ότι αυτές οι θέσεις εργασίας που έχουν ε, το χαρακτηριστική ονομασία Mac Jobs είναι θέσεις απασχόλησης ε, υποδέστερες ας πούμε που δεν χρειάζονται μεγάλη εξειδίκευση και εργάζονται κυρίως φοιτητές ε, Στόχο είναι όμω να μετακπαιδευτούν και να επασχοληθούν αλλού. Ε, και σε ό,τι αφορά τη μετακπαίδευση και την κατάρτιση εργαζομένων στο εσωτερικό τη εταιρεία, ε, το κόστος το επομίστηκε σχεδόν 100% η ίδια εταιρεία McDonald's. Και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φροντίσουν και οι ίδιοι να προάγουν τα προσόντα τους και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να γίνεται καμία διάκριση για το πού ε, απασχολούνται οι εργαζόμενοι. Ο στόχος θα πρέπει να είναι πάντα ο ίδιος. Η εκάστοτε αναβάθμιση των προσόντων της ποιότητάς τους για τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Και επειδή ε, η αγορά εργασίας, ε, ο κόσμος της εργασίας είναι κάτι που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη κινητικότητα, να μην είναι εκτεθειμένη στην ανεργία. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα λοιπόν στην ε, ερώτηση των υπαριθμών 16 σχετικά με το μέσο μικροχρηματοδότηση ευρωπαϊκής πρόοδου. Επίτροπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω τη χαρά να σας πω ότι ε, και τα δύο αυτού του προγράμματος και το τμήμα των εγγύσεων και το τμήμα της ρευστότητα και τα δύο αυτά λειτουργούν. Ε, τρεις μήνες μετά τη θέση σε ισχύ της απόφασης η Κομισιόν ε, ολοκλήρωσε την εντολή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ε, να προσφέρει τις εγγύσεις. Το Νοέμβρη η Κομισιόν συνέστησε ένα ειδικό εργαλείο επενδύσεων και κατόπιν τούτου οι πρώτες μικροχρηματοδοτήσεις, τα μικροπιστώσεις θα δίδονται από αυτό το μήνα. Και με μεγάλη μου χαρά μπορώ να σας πω ότι η Κομισιόν κατόρθωσε να διασφαλίσει ε, και περαιτέρω χρηματοδότηση σε ε, μικροεπιχειρηματίες. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συνεισφέρει και αυτή 100 εκατομμύρια ευρώ ε, και αναμένεται να συνεισφέρουν και άλλοι. Κατόπιν τούτου το σύνολο των πιστώσεων θα αυξηθεί σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Ε, τα χρήματα αυτά θα ωφελήσουν τους ανέργους όσο αντιμετωπίζουν τον αποκλεισμό ή ευάλωτα άτομα που έχουν δυσκολία ε, στο να μπουν στην αγορά. Μας ενδιαφέρει λοιπόν αυτή η ομάδα, η, μας ενδιαφέρει και η γεωγραφική ισορροπία και αυτά είναι καθοριστικά στοιχεία της εντολής που έδωσε η Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μέχρι τώρα προετοιμάζονται συγκεκριμένε δράσεις έτσι ώστε να ε, επιτευθούν και οι δύο στόχοι. Από τις αρχές του 2011 οι μικροπιστώσεις ε, θα αρχίσουν να χορηγούνται ε, κυρίως στο Βέλγιο για να αντιμετωπιστούν μειονεκτούς περιοχές αλλά και στην Ολλανδία σε άτομα που δεν έχουν καμία πρόσβαση σε συμβατική χρηματοδότηση. Η όλη αυτή η λειτουργία ε, θα είναι ισόρροπη, όπως σας είπα θα καλύπτεται και το γεωγραφικό στοιχείο. Θεωρώ ότι πάνω από 40% ε, θα δοθούν ε, στην κεντρική Ευρώπη. Είναι γνωστό ότι οι μικρο επενδύσεις είναι πιο αποτελεσματικές και όταν συνοδεύονται από υπηρεσίες στήριξης. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει μέτρα ε, για να στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αλλά και όλους τους άλλους ε, για να ε, <clears throat> στηριχθεί η αυτοαπασχόληση και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα κράτη-μέλη έχουν πάρει πάνω από 2,7 δις ευρώ ε, οι επιχειρηματίες μπορούν και αυτοί να στηριχθούν. Βέβαια κατά πόσον ε, τα επιτόκια θα επιδοτούνται. Αυτό είναι μια απόφαση ε, που πρέπει να λαμβάνει το ίδιο το κράτος μέλος. Μέχρι τώρα μόνο η Λιθουανία έχει αναφέρει ότι θα κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας. Και τέλος η Κομισιόν θα δώσει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο αυτού του εργαλείου των μικροπιστώσεων. Ε, θα προσφέρουμε επίσης πληροφορίες για αυτές τις μικροπιστώσεις. Η Κομισιόν θα χρησιμοποιήσει τα υπάρχοντα δίκτυα της ε, ε, απασχόλησης. Ε, οι ΜΚΟ και άλλοι φορείς ε, καλούνται να προσφέρουν πληροφορίες για την πρόοδο αυτών των επιστώσεων. Εξάλλου θα αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία και στους νέους με διαφορετικά προσόντα για να μπορούν και αυτοί να ξεκινήσουν τη δική τους τη δουλειά και να λάβουν μικροπιστώσεις. Ευχαριστώ. Κύριε επιστρέψουμε μετά στην ερώτησή σας στη 15, μετά την διεκπαιρέωση της 16ης ερώτησης. Έχω μία συμπληρωματική για το θέμα αυτό. Ναι, αλλά έχουμε ήδη τρεις συγγραμμένες και συμπληρωματικές. Την κυρία Γκέντς, τον κύριο Ζέμ, και την κυρία Τσικάου. Αργότερα θα ακούσουμε τη δική σας ερώτηση. Κυρία Γκέντς. Ευχαριστώ. Χαίρομαι. Χαίρομαι για την απάντηση που μας έδωσε ο Επίτροπος. Πριν από λίγες εβδομάδες λάβαμε μία έκθεση του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου που ανέφερε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ή κάτι τέτοιο. Αρχικά 500 εκατομμύρια ευρώ είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό για το μέσο μικροχρηματοδότησης γιατί χρειάστηκαν συμπληρωματικοί πόροι, γιατί χρειαζόμαστε το πρόγραμμα αυτό για να μετριάσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν μπορεί να δώσει επιδοτήσεις ε, για κατάρτιση ή επιμόρφωση. Γιατί αυτή ήταν, αυτός ήταν ο αρχικός προορισμός και ο στόχος του ΕΚΤ. Φαίνεται όμως ότι αμελήθηκε στην πορεία. Και να δώσουμε έμφαση σε αυτούς που χρειάζονται περισσότερο τέτοιου είδους προγράμματα. Είναι πιο ευάλωτοι. Θα ήθελα κύριε Επιτρόπε, να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Συμφωνώ απόλυτα ότι το μέσο αυτό, το μέσο μικροχρηματοδότησης, είναι πολύ σημαντικό και αξιόλογο. Θα πρέπει όμω ε, να έχουμε υπόψη ότι θα πρέπει να απαντήσουμε και στην ερώτηση ποιες χώρες αξιοποιούν το μέσο μικροχρηματοδότησης. Με ανησύχησε ένα στοιχείο της απάντησης, της σας που είπατε ότι υπάρχει διαφοροποίηση και γεωγραφική και εθνική. Θα, θέλετε, θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι οι χώρες που αξιοποιούν περισσότερο αυτό το μέσο μικροχρηματοδότηση. Κυρία Τσικάου, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μισό λεπτό. Κύριε Επιτροπέ, σίγουρα οι νέοι είναι οι πιο ευάλωτοι απέναντι στην κρίση και έχουν πληγεί περισσότερο από αυτήν, αλλά θα πρέπει να ξεχνούμε και τους α, ε, άνω των 40 ετών που είναι άνεργοι. Αναφέρατε ότι το 60% του μέσου μικροχρηματοδότησης ε, θα κατευθυνθεί προς χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης διαπιστώσατε φραγμούς που εμποδίζουν τη χρήση του μέσου μικροχρηματοδότησης σε αυτή ακριβώς ε, τη γεωγραφική περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που δείξατε, για το θέμα των μικροπιστώσεων, για το θέμα αυτό ε, πράγματι ε, είναι ένα θέμα που εξετάζεται από διάφορες γενικές διευθύνσεις. έχει σχέση και με την περιφερειακή πολιτική και εκεί ασχολούμεθα με το θέμα αυτό. Όσον αφορά τα επιτόκια, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένα κρατημέλη τα οποία βάζουν ως προϋπόθεση ένα ανώτατο όριο το οποίο βρίσκεται περίπου σε 8 με 9,5%. Βεβαίως ε, θα πρέπει να έχει κανείς κατά νου ότι και αυτό ήταν ένα θέμα κατά την προετοιμασία του θέματος να έχει κανείς κατά νου ότι τα πάγια έξοδα είναι αρκετά υψηλά σε σχέση με ε, τις πιστώσεις. Πρέπει λοιπόν να καλυφθούν αυτά τα έξοδα, πρέπει να αναστηθεί ε, μια μεσαίωδος και νομίζω το καταφέραμε αυτό. Όσον αφορά το άλλο σας ερώτημα, μπορώ να σας πω ότι με το εργαλείο Jasmine έχουμε ως στόχο να προετοιμάσουμε τη μικροκρηματοδότηση, να προετοιμάσουμε τους ε, ενδιάμεσους. Αυτή τη στιγμή έχουμε 15 θεσμούς ε, που προετοιμάζουν 15 οργανισμούς σε 15 ε, διαφορετικές χώρες. 11 βρίσκονται στην κεντρική στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τέσσερις ε, στη Δυτική Ευρώπη. Ε, βέβαια δεν έχω κατά νου όλες αυτές τις ε, χώρες αλλά πρόκειται κυρίως για τις ε, νέες χώρες και υπολογίζουμε ότι κατά τα επόμενα έτη θα προσθεθούν και άλλες 20 ενδιάμεση μέσω του προγράμματος Jasmine. Ε, για το τελευταίο ερώτημα, ε, παρακαλώ να δείξετε κατανόηση. Δεν μπορώ να σας ε, δώσω αυτή τη στιγμή απάντηση. Θα σας απαντήσουμε γραπτά και θα αναφερθούν λεπτομερώς τα αίτια, οι λόγοι γιατί υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στην πρόσβαση. Ε, πολλές φορές βέβαια υπάρχουν και προβλήματα επικοινωνίας. Υπάρχουν εμπόδια, κυρίως όταν ε, πολλοί από τους ε, δυνάμει πιστολήπτες είναι εκείνοι οι οποίοι δεν θα παίρναν δάνειο και από μια κανονική τράπεζα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει κάποια επιφύλαξη. Υπάρχει επιφύλαξη ως εκ τούτου είναι απαραίτητο στον τομέα αυτό να υπάρξουν περαιτέρω Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον Επίτροπο και πάμε τώρα στην ε, ερώτηση υπαριθμών 15 του κυρίου Μπαλτσίτης. Επίτροπος Ταγιάννη, που θα απαντήσει. Signor Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτέ. ο ευρωπαϊκός κλάδος του τουρισμού, όπως και πολλοί άλλοι οικονομικοί τομείς, ε, καλείται να αντιμετωπίσει μια μεγάλη πρόκληση, την πρόκληση της ε, παγκοσμιοποίηση. Ε, πρόκειται για μια πρόκληση όπου η Κομισιόν έχει αναφερεί και έχει τοποθετηθεί κυρίως με την ανακοίνωσή της που έχει εκδώσει ε, στις 30 Ιουνίου του περασμένου έτους. Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει και μια ειδική ανακοίνωση για τον τουρισμό όπου προτείνεται μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική, η στρατηγική του 2020, μια σταθερή πολιτική για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ε, τομέα. Να υπάρχει λοιπόν μια ε, σταθερή πολιτική. Έχουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα και αυτό είναι μια θεμελιώδης αρχή της σταθεροποίησης. Ε, το να επιτύχουμε βέβαια το στόχο, για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να προκαλέσουμε την ανταγωνιστικότητα στον ε, τομέα του τουρισμού. Δεύτερον, να ε, στηρίξουμε έναν τουρισμό μεγάλης διάρκειας και κατόπιν να σταθεροποιήσουμε την εικόνα και την παρουσία της Ευρώπης ε, ως στόχο των τουριστών, ως τουριστικό στόχο και πρέπει βεβαίως και να βελτιστοποιήσουμε τα εργαλεία που υπάρχουν για να αναπτυχθεί περαιτέρω ο τουρισμός. Οι πρωτοβουλίες ε, θα πρέπει να αποδώσουν στον τομέα τα εργαλεία για να προσαρμοστεί στις ε, προκλήσεις και στόχος όπως είπαμε είναι να υπάρχει τουρισμός διάρκειας και ανταγωνιστικός. Βεβαίως και είναι απαραίτητο να ληφθούν και συγκεκριμένα μέτρα να βελτιωθεί η ποιότητα των παραχώμενων τουριστικών υπηρεσιών και να βελτιωθούν ε, οι δεξιότητες ε, των απασχολούμενων στον τουρισμό. Γιατί δεν μπορούμε πλέον να σκεπτόμεθα τον τουρισμό ως ε, ένα τομέα που είναι οικογενειακή υπόθεση, ε, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ε, ένα πιο σύγχρονο ε, τουρισμό, ανταγωνιστικό. Και θα σας αναφέρω και κάποια παραδείγματα όσον αφορά την εκπαίδευση των απασχολούμενων. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο έχει και άμεση σχέση και με τις νέες τεχνολογίες για να υπάρχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Αυτές είναι προτάσεις οι οποίες έχουν μπει στο κείμενο Τη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα κείμενο το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο. Ε, ένα κείμενο ε, το οποίο έχει συζητηθεί και στο Κοινοβούλιο. Η κινητοποίηση λοιπόν των παραγόντων του τουρισμού για την βέλτιστη χρήση των προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα Λεωνάρντο, ένα πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα, έρασμους ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλα προγράμματα. Να υπάρχει και μια στρατηγική για την τουριστική προσφορά που θα είναι διαφορεποιημένη αυτή να υπάρχει ηλεκτρονική υποστήριξη για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Αυτά θα επιτρέψουν να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για τους ε, παράγοντες του κλάδου. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να υποφεληθούν και από άλλες οριζόντιες πρωτοβουλίες για πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Και εδώ αναφέρομαι στην περίπτωση Jeremy, μια πρωτοβουλία που κινούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για βελτιωθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως μέσα από ε, κεφάλαιο κινδύνου, μικροπιστώσεις και άλλες μορφές ε, ενισχύσεων. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τουρισμό, οι επιχειρήσεις αυτές επωφελούνται πλήρως από τα μέτρα που έχουν ε, προταθεί κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Κοινοβούλιο θα λάβει το επικαιροποιημένο κείμενο μετά από λίγες μόνο εβδομάδες. Έτσι λοιπόν και αυτό είναι ένα εργαλείο για να προστατευτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού οι οποίες αποτελούν μια τεράστια δύναμη για να αναπτυχθεί περαιτέρω ένας τομέας σημαντικός για μας κατά τα επόμενα έτη γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι μια ευρωπαϊκή πολιτική όπως προβλέπεται από τη συνθήκη θα αποφέρει προστιθέμενη αξία ε, σε ε, δουλειά ε, την οποία κάνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι μπορώ να διαβεβαιώσω τον αξιότιμο κύριο βουλευτή που υπέβαλε αυτή την ερώτηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι συνεργάτες μου θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να έχουν πρόσβαση στα κοινοτικά μέσα χρηματοδότησης και αυτά στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που έχει ως στόχο ο τουρισμός να είναι κομβική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Βαλτσίτης και μετά άλλοι ομιλητές, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνάδελφο Μπαλτσίτης. Πρώτα εσείς, ε, ο κύριος Μπαλτσίτης μετά εσείς και μετά κυρία Τσικάου, παρεξήγηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριος Μπαλτσίτης. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εκτενέστατη απάντησή σας Όλοι όσοι σας άκουσαν ελπίζουν τα όσα είπατε για την ανάπτυξη του τουρισμού να γίνουν πραγματικότητα στο μέλλον και να είναι ε, ελκυστικός και αυτός ο τομέας για επενδύσεις. Όπως γνωρίζετε, η τουριστική βιομηχανία δεν γνωρίζει ε, την ίδια ανάπτυξη στην Ευρώπη για λόγους υποκειμενικούς όσο και αντικειμενικούς. Έχουμε μια στρατηγική για τη Βαλτική και η ελκυστικότητα της ε, περιοχής της Βαλτικής είναι ένα από τα στοιχεία αυτά και μάλιστα πρωτοαρχικός στόχος. Τι έχουν γίνει στον τομέα ε, αυτό, ποια είναι τα επιτεύγματα τα τελευταία χρόνια. Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη που διακόψα προηγουμένω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Μπαλτσίτη για αυτή την ερώτηση, η οποία ε, φέρνει στο επίκεντρο αυτό το επιχείρημα, το οποίο θα κληθεί το Κοινοβούλιο να αντιμετωπίσει και κατά του επόμενου ε, μήνε. Ε, γιατί έχω μια εισήγηση από αυτού να πω στον κύριο Ταγιάννη ότι πράγματι έδωσε όθηση στον ε, τουρισμό ε, και με βάση τα αρμοδιότητες ε, που προβλέπουν οι συνθήκη τη Λισαβόνα. Είχαμε μία ανακοίνωση τον προηγούμενο Ιούνιο και την παρουσίαση προγράμματο. παρουσιάστηκε πριν από λίγε μόνο εβδομάδες. Αυτά τα δύο έχουν ω επίκεντρο την προσοχή στι μικρομεσαίες επιχειρήσει να γίνουν πιο ανταγωνιστικέ. Καινοτομία, εκπαίδευση, βασικά στοιχεία. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση υπάρχουν εδώ δύο σημαντικά θέματα. Πρώτον, να γίνεται καλύτερη χρήση. Μισό λεπτό, λέει ο πρόεδρο. Μισό λεπτό. Διακόπτη, αλλά γελάει ο πρόεδρος γιατί μιλάει με απίθανη ταχύτητα, ασύλληπτη ταχύτητα ο μιλητή. 30 δευτερόλεπτα για τη συμπληρωματική ερώτηση, κυρία Τσεκάου. Ευχαριστώ πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε. Ορισμένες χώρες χρησιμοποιούν τα περιφερειακά προγράμματα για την ε, ανάπτυξη και τη γενοτομία. Επί παραδειγμή το Ηνωμένο Βασίλειο ή και η Ελλάδα και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν σκέφτεστε να δημιουργήσετε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για να βελτιωθεί η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση για τον τουρισμό συγκεκριμένα. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε.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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαλτσίτης γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να παρέμβω ε, σε ένα θέμα που το έχω ενστερνιστεί ε, και για το οποίο βέβαια είμαι και αρμόδιος ε, για τον τουρισμό. Επειδή είμαι ο πρώτος επίτροπος αρμόδιος για τον τουρισμό θεωρώ πράγματι ότι αυτό το θέμα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το θέμα είναι θέμα κλειδί. Αλλά για να απαντήσω πιο συγκεκριμένα πέρα από τις πολιτικές πρωτοβουλίες που Προσπάθησα να υλοποιήσω από τότε που έγινε επίτροπος και τα είπε και αυτό και ο κύριος ε, Φιντάντσα. Γιατί εδώ ε, η πολιτική του τουρισμού πριν από τις συνθήκες Λισαβόνας δεν ήταν ε, κοινοτική αρμοδιότητα. Άρα δηλαδή δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια για να συμβάλλουμε σε μια σημαντική ε, κοινοτική δράση. Έχουμε προγράμματα ενδιαφέροντα όπως το πρόγραμμα Καλυψό που αξιολογήθηκε στην Ισπανία. Αλλά αν κατάλαβα καλά, το μήνυμα που πέρασε ο κύριος Φιντάντσα στην έκθεση που θα παρουσιάσει το Κοινοβούλιο, εκεί θα αναφέρεται υποστήριξη ε, της αυξήσης ε, των κονδυλίων για τον ε, τουρισμό. Αυτό μπορεί να συμπεριληφθεί στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο, ad hoc. Είναι όμως σημαντικό το Κοινοβούλιο να επιληφθεί του θέματος, γιατί είναι δύσκολο να δώσει κανείς συγκεκριμένες απαντήσεις αν δεν υπάρχουν τα οικονομικά εργαλεία. Τούτο βέβαια δεν σημαίνει ότι και εμείς δεν θα κινηθούμε αποφασιστικά. Οι ε, πρωτοβουλίες είναι πάρα πολλές, αυτές που έχουν αναλυφθεί. Η Βελγική Προεδρία έχει οργανώσει, οργάνωσε μια μεγάλη εκδήλωση στη Μάλτα. Ε, το ίδιο είπε και η Ουγγρική Προεδρία. Μας το είπε αυτό πριν από λίγες μέρες όταν συναντηθήκαμε στη Βουδαπέστη. Θα οργανώσει μια μεγάλη εκδήλωση με αντικείμενο τον τουρισμό. Είμαι ικανοποιημένος από ε, συνάδελφος κ. Μπαλτσίτης ε, έθιξε και το θέμα του τουρισμού στη Βαλτική γιατί ο τουρισμός δεν αφορά μόνο τη Μεσόγειο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Μάλτα. Ο τουρισμός είναι σημαντικός πόρος για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της ε, Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης που έχουν ομορφιές και που μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω. Όσον αφορά τις χώρες της Βαλτικής, θεωρώ ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζεται στο κείμενο που εγκρίθηκε στις 30 Ιουνίου του περασμένου έτος είναι η σχέση με την αναδυόμενη νέα αστική τάξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας όπου υπάρχουν εκατομμύρια πολιτών και ε, θέλουν να ε, ταξιδέψουν. Αυτοί ε, θέλουν να βγουν από τα σύνορα της χώρας τους. Έχουμε πρόβλημα με τις θεωρήσεις, το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με την Κίνα και νομίζω ότι οι Υπουργοί Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα για να εκμεταλλευτούν τους Ρώσους τουρίστες το τους δυνάμει τουρίστες και τους Κινέζους έτσι ώστε να είναι πολύ πιο εύκολο να τους δεχτούμε αυτούς ε, στις χώρες μας και επειδή οι χώρες Βαλτικής είναι πιο κοντά στη Ρωσία αυτές μπορούν να υποφαληθούν καλύτερα από αυτή την αναδυόμενη αστική τάξη της Ρωσίας που θα φέρει πολλά χρήματα στη Βαλτική. Αυτά λοιπόν μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα ε, όσον αφορά τις ε, τουριστικές ε, δραστηριότητες. Χαίρομαι που πολλοί υπουργοί από διάφορες χώρες συνάντησαν πριν από κάποιες εβδομάδες στο Λονδίνο το νέο Βρετανό Υπουργό Τουρισμού. Και η Μεγάλη Βρετανία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να στηρίξει την τουριστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το και η Γαλλία. Είναι λοιπόν σημαντικό να βρούμε και κάποιες πύλες εισόδου. Γιατί η Ευρώπη ε, πρέπει να προσφέρει προστιθέμενη αξία και χαίρομαι που η κυρία Βασιλείου ε, έχει και αυτή τη δική της συνεισφορά στον αθλητισμό, ας πούμε στο Λονδίνο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι μοναδική ευκαιρία για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρέπει κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πύλη εισόδου, να μπαίνουν εκεί οι τυρίστες, να μην μένουν εκεί, αφού επισκεφτούν από τη χώρα να πηγαίνουν και σε άλλες ευρωπαϊκές. Αυτή είναι μια κοινή δράση ε, που αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ είναι καθοριστική σημαντική η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για όλα αυτά που προσφέρετε ε, στη συζήτηση για τον τουρισμό αλλά και για όλες τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν ε, στο μέλλον για τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και προχωρούμε τώρα στις ερωτήσεις προς την κυρία Βασιλείου. Η πρώτη είναι της κυρίας Μπλίνκεβιτσούτε με θέμα, όποτε είστε έτοιμοι κύριε Επίτροπη, πρωτοβουλίε και προγράμματα εξυγχρονισμού τη ανώτατη εκπαίδευση. Ερώτηση παριθμό 17. Είστε έτοιμοι κύριε Βασιλείο, έχετε το λόγο, όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η εκπαίδευση είναι από τους βασικούς παράγοντες ε, που ευνοούν την απασχολησιμότητα οι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης έχουν 40% λιγότερες πιθανότητες να είναι άνεργοι. Ωστόσο, η υποαπασχόληση και η ανεργία των νέων είναι υπερβολική σήμερα. Πάρα πολλοί πτυχιούχοι αγωνίζονται να περάσουν στην αγορά εργασίας και να έχουν μια ασφαλή θέση απασχόλησης που να ανταποκρίνεται και ε, την εκπαίδευσή τους και στη μόρφωσή τους. Βεβαίως τα προβλήματα και τα θέματα ξεκινούν πολύ πριν την ανώτατη εκπαίδευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για να εντοπίσει τις βασικές ικανότητες όσο και δεξιότητες που θα πρέπει να ε, μαθαίνουν να αποκτούν οι νέοι στο σχολείο. Θα σήμερα καλούνται οι νέοι να έχουν πολύ περισσότερα προσόντα από ό,τι ποτέ στο παρελθόν για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να ανθίσουν σε μια παγκόσμια οικονομία και πολλοί θα χρειαστεί να απασχοληθούν σε θέσεις απασχόλησης, σε δουλειές που δεν υπάρχουν ακόμα. Η μεγάλη ε, δυνατότητα και ε, γλωσσικές ικανότητες και ικανότητες προσαρμογής σε ένα κόσμο πολυπολιτισμικό. Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο με τρόπους που ούτε καν διανοούμαστε. Δηλαδή η δυνατότητά τους να συνεχίσουν να διδάσκονται, να μαθαίνουν και να καινοτομούν θα είναι σημαντικοί παράγοντες για την απασχολησιμότητά τους. Έχει σημασία και η καθοδήγηση των νέων. Οι νέοι όλο και περισσότερες επιλογές έχουν στη διάθεσή τους για την εκπαίδευσή τους. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις με τα λόγου γνώση αυτό σημαίνει και απαιτεί καλύτερη εκπαίδευση για τη μόρφωσή τους, καλύτερη ενημέρωση για την εκπαίδευση, για την κατάρτιση, για τις θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ποιοτικό επαγγελματικός προσανατολισμός, με ποιότητα, με μεγάλη συμμετοχή και τη ίδια της αγοράς και των θεσμών της. Έρχομαι τώρα στην ανώτατη εκπαίδευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα, όπως γνωρίζετε, ε, είχε μια βληματική πρωτοβουλία νεολαία σε κίνηση για το 2020 για να είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση ε, πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες των νέων. Τώρα ερχόμαστε στην ε, εφαρμογή, υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του 2011, θα ε, έχουμε μια νέα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εξυγχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης. Θα καταγράψουμε τις προόδους που έχουν γίνει για να είναι πιο προσαρμοσμένοι στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας που βασίζεται στη γνώση. Και εδώ συμπεριλαμβάνεται και το θέμα της απασχολησιμότητας. Θα εντοπίσουμε τις βασικές προκλήσεις για το μέλλον και θα εκπονήσουμε την απάντησή μας. Τμήμα λοιπόν αυτών των προσπαθειών μας είναι και η ευρωπαϊκή πλατφόρμα που θέλουμε να ενισχύσουμε για το διάλογο μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων για να αυξάνεται η απασχολησιμότητα των φοιτητών και να έχει μεγαλύτερο ρόλο η ανώτατη εκπαίδευση στο τρίγωνο της απασχόλησης. Χρειάζεται διαφάνεια σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Για τον τρόπο με τον οποίο παρέχουν τη μόρφωση τα ανώτατα ιδρύματα, αυτό ενισχύει και τη συνεργασία αλλά και τον ανταγωνισμό των πανεπιστημίων την άμυλα για να βελτιωθεί η συνεργασία τους. Υπάρχουν διεθνείς βαθμολογίες σήμερα των πανεπιστημίων, αλλά δεν δίνουν πλήρη εικόνα των επιδόσεων των, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα μιας μελέτης σκοπιμότητας για να δούμε ένα εναλλακτικό σύστημα βαθμολόγηση των πανεπιστημίων, ένα πολύπλευρο που θα αντικατοπρίζει τη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία των πανεπιστημίων. Θα πρέπει καλύτερα να προλαμβάνει η Ευρώπη να προβλέπει τις ικανότητες και δεξιότητες που θα χρειάζονται οι νέοι μας στο μέλλον. Γι' αυτό προωθεί και μια νέα ατζέντα που συνδυάζεται χέρι-χέρι με την πρωτοβουλία μας για την νεολαία κίνηση. Να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους μας να βρίσκουν ε, πιο εύκολα δουλειά να έχουν το σωστό μείγμα δεξιοτήτων, ικανοτήτων, να προσαρμόζονται σε μια κοινωνία που αλλάζει με ταχύς ρυθμούς. Είναι ένα νέο πανόραμα που θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2011 για να μπορέσουμε να προβλέπουμε όχι μόνο τις ικανότητες που θέλουν σήμερα οι εργοδότες αλλά και αυτές ε, και τα προσόντα που θα ζητούν στο μέλλον. Φέτος λοιπόν την Άνοιξη προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέες ευρωπαϊκές ε, μορφές αξιολόγησης, κριτήρια, benchmarks για να μπορούν οι νέοι στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας που βασίζεται στη γνώση να βρίσκουν δουλειά. Επίσης, προγράμματα για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας και προγράμματα ανταλλαγής ε, φοιτητών και μετακίνησης τύπου Εράσμους θα βελτιώσουν τις ευκαιρίες που έχουν οι νέοι να βρίσκουν δουλειά γιατί αποκομίζουν πολύτιμη διεθνή εμπειρία και ε, προάγουν και τις διανοητικές τους ικανότητες και τον νου τους. Ευχαριστώ. δεύτερα παρακαλώ Μπλίνκεβιτσούτε, Ζέμκα και Παπα-Νικολάου. Με αυτή τη σειρά. Πρώτα κυρία Μπλίνκεβιτσούτε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Ήταν πολύ εκτενής ε, η απάντησή σας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εγγυάται το δικαίωμα στην ποιοτική εκπαίδευση σε όλους τους πολίτες. Υπάρχουν όμως μεγάλες διαφορές μεταξύ των ανωτάτων ιδρυμάτων ε, των διαφόρων κρατών μελών. Ε, υπάρχουν διάφορα συστήματα χρηματοδότησης, ε, δανειοδότησης των φοιτητών υποτροφιών. Όταν παίρνουν δάνεια φοιτητέ είναι πάρα πολύ ψηλά όμως τα επιτόκια και πάρα πολύ επαχθείς οι όροι αποπληρωμής. Και αυτό αποθαρρύνει τους φοιτητές και φεύγουν από τις χώρες μας και πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Διαρροή εγκεφάλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτείνει. δεν Θα κάνει τίποτα γι' αυτό, για τα φοιτητικά δάνεια. Ο κύριος Ζέμκε, έχω μία ερώτηση μόνο, γιατί θα μπορούσαμε να επεκταθούμε σε πολλά θέματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Επίτροπε, ε, συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διευρυθούν οι πόροι των προγραμμάτων σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή νέων στην Ευρώπη. Γιατί έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια... Ε, τα κονδύλια που έχουμε για το έρασμο ή για άλλα προγράμματα είναι, ε, μένουν μετακίνητα και οι υποτροφή είναι πολύ χαμηλέ. Δεν υπάρχει καμία αύξηση των κονδύλιων τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ. Κύριε Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ κύριε, ε, κύριε Πρόεδρε. Είναι αλήθεια, κυρία Επίτροπε, πω το συγκεκριμένο ζήτημα εμπίπτει σε θέματα επικουρικότητο. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πόρου για τον εξυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών των κρατών μελών για παράδειγμα θυμίζω ότι στο προηγούμενο το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη πολλά κράτη μέλη απορρόφησαν κοινοτικού πόρου για αυτό το σκοπό και το ερώτημα είναι συγκεκριμένο διαθέτει η επιτροπή στοιχεία για την αποτελεσματικότητα αυτών των πόρων που δόθηκαν αλλά και θα δοθούν στα κράτη μέλη. Η κυρία Βασιλείου, καταρχάς για το θέμα των διαφορών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των πανεπιστημίων ακριβώς περί αυτού πρόκειται και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε διαφάνεια ε, τις επιδόσεις των πανεπιστημίων. Γι' αυτό ολοκληρώνουμε τώρα τη μελέτη αντικτύπου, σκοπιμότητας μάλλον, για να δούμε πώς θα βαθμολογηθούν τα πανεπιστήμια, θα έχουμε και μια χαρτογράφηση των πανεπιστημίων με προδιαγραφές, στάνταρ, κριτήρια, έτσι ώστε οι φοιτητέ να είναι πιο ενημερωμένοι στην επιλογή τους και να ξέρουν ακριβώς πού να πάνε να σπουδάσουν, τι να σπουδάσουν και τι παρέχει το πανεπιστήμιο και τι προδιαγραφές έχει αυτό το οποίο θέλουν να εισαχθούν. Σε ό,τι αφορά τα δίδακτρα έχετε δίκιο. Όταν υψηλά τα δίδακτρα πρέπει να είναι και δίκαια τα δάνεια τα φοιτητικά. Αλλά όπως γνωρίζετε βεβαίως αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι συμφωνούν οι οικονομολόγοι ότι η επένδυση στην εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Ε, πάντα λοιπόν εγώ καλώ τις κυβερνήσεις να μην κάνουν περικοπές στις επενδύσεις στην παιδεία ή στα πανεπιστήμια. Επιπλέον, συμφωνώ με το αξιότιμο μέλος που έκανε την ερώτηση αυτή για την ανεπάρκεια των ε, δανείων ε, για προγράμματα κινητικότητας ανταλλαγής φοιτητών, όπως είναι ο Έρασμος. Γι' αυτό και πάλι θα ε, γίνει μια μελέτη, ελπίζω να ολοκληρωθεί σύντομα, μελέτη της London School of Economics, που διερευνούμε τη δυνατότητα που έχουν τα όργανα της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό φοιτητικό δάνειο για την κινητικότητα των φοιτητών. Αυτό είμαι βέβαια θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές, είτε είναι φτωχοί είτε είναι πλούσιοι, να μπορούν να ταξιδεύουν, να μετακινούνται και να υποφελούνται αυτών των προγραμμάτων και των δανείων. Για τον κύριο Παπα-Νικολάου τώρα και την ερώτησή του. Μιλά για τα διαρθρωτικά ταμεία, ε, για την ανάπτυξη ε, βάσει των οποίων μπορούν τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν την υποδομή τους για την παιδεία. Δυστυχώς, ακριβώς όμως επειδή δεν είναι δική μου αρμοδιότητα τα διαρθρωτικά ταμεία, δεν ξέρω, θα ρωτήσω τον κύριο Χάν εάν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, εάν υπάρχουν τέτοιες εκθέσεις ως προς το αποτέλεσμα των ε, δανείων και θα σας ενημερώσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και ερχόμαστε τώρα στην ώρα της κυρίας ε, ε, Mork United για τις μαθητικές επιδόσεις στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ, κυρία Πέτροπα, έχετε το λόγο. Thank you, President. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως θα γνωρίζετε, κάθε κράτος μέλος αποφασίζει πώς θα οργανώσει το εκπαιδευτικό του σύστημα. Αυτό αφορά το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνάδει με αυτό. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για να προωθήσει την αμοιβαία εκμάθηση και την ανταλλαγή βέλτιση των πρακτικών. Όπως είπαμε και στη στρατηγική για την Ευρώπη το 2020 είναι ζωτικό για το μέλλον της Ευρώπης που θα είναι μια κοινωνία που θα στηρίζεται στη γνώση να εξυγχρονίσει τα εκπαιδευτικά της συστήματα προκειμένου να έχει τα πιο προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο. Και μάλιστα οι μελέτες του ΩΣΑ είναι σημαντικές ε, για, ε, για τον απολογισμό αυτών των, προσ, ε, προσπαθειών. Και μάλιστα η τελευταία μελέτη πίσα του ΩΣΑ του 2009 δείχνει κάποια στοιχεία βελτίωσης σε ορισμένους τομείς, αλλά ε, επισημαίνει ότι πολλή πρόοδος θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη και αυτές οι μελέτες ε, δίνουν ε, σημαντικές πληροφορίες και στα κρατημέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Συγκριτικός Κανόνας που υθέτησε το Συμβούλιο το Μάιο του 2009 έχει στόχο τις βασικές δεξιότητες στην ανάγνωση, μαθηματικά και επιστήμες και μάλιστα Θέλουμε να βελτιωθούν οι μαθητικές επιδόσεις για μαθητές κάτω των 15 μέχρι το 2020. Θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι από την μελέτη PISA που είναι πολύ εύστοχο. Και μάλιστα το μερίδιο των χαμηλών επιδόσεων μαθητών στην ανάγνωση που είχε αυξηθεί από 21% το 2000 σε 24% το 2006 βελτιώθηκε, πέρασε στο 20% το 2009. Βέβαια, ο συγκριτικό κανόνας για το 2010 προκειμένου να μειώσουμε το 20% στο 17% δεν έχει υλοποιηθεί δυστυχώς. Σε ό,τι αφορά τη, τα μαθηματικά και τις επιστήμες είχαμε μείωση το 2006, είχαμε περισσότερη πρόοδο στην επιστήμη από στα μαθηματικά και το μερίδιο των κακών μαθητών είναι σήμερα χαμηλότερο στις επιστήμες από ό,τι στα μαθηματικά. Τώρα, αν το 2006 χρησιμοποιηθεί ως ε, σημαντικό σημείο αφετηρίας, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει σε καλό δρόμο για την πρόοδο που θέλει να, σημειώσει μέχρι το 2020 σε ό,τι αφορά το συγκριτικό κανόνα για τους ε, κακούς μαθητές. Πάντως, ε, στις 25 χώρες για τις οποίες έχουμε στοιχεία φαίνεται ότι 22,5% των κακών μαθητών είχαμε το 2006 και μέχρι το 2009 το μερίδιό τους ε, μειώθηκε στο 19,6% το μερίδιο των κακών μαθητών. Δηλαδή, κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε κάποια πρόοδο ό,τι αφορά τον περιορισμό των κακών μαθητών. Βέβαια, θα εξετάσουμε τα αποτελέσματα της ε, μελέτης PISA και θα δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματά μας και τα συμπεράσματά μας τον έβριο του 2011. Πάντως, ε, προσκαλέσαμε τα κράτη-μέλη να επικεντρωθούν στους ε, εξή τομεί. Να δώσουμε κίνητρα για τη βελτίωση στην ανάγνωση, μαθηματικά, νέες τεχνολογίες, ε, επίπτωση νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, προκειμένου να αποκτήσουν αυτονομία οι μαθητές και να έχουν όλο και περισσότερα κίνητρα, βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, ε, και θέματα καθηγητών εκπαίδευση, επιμόρφωση καθηγητών και θέματα διοντολογικά για το σχολείο και τα χαρακτηριστικά του. Επίση, στα συμπεράσματα του, το Συμβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ιδρύσει μια ομάδα υψηλού επίπεδου για, την, ε, για τα μαθηματικά, τη τεχνολογία και τα μαθηματικά και ένα για την ανάγνωση. Και μάλιστα θα ξεκινήσει τι από την 1η Φεβρουαρίου. Θα ασχοληθεί με τα μέτρα καλών βέλτιστων πρακτικών στην έρευνα και στις, ε, στην προσπάθεια των κρατών μελών να βελτιώσουν ε, την, ε, τις στρατηγικές διαβίου κατάρτισης ό,τι αφορά την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων. Μάλιστα η ομάδα αυτή θα ολοκληρώσει το έργο της και θα δημοσιεύσει τις, τα συμπεράσματά της στα μέσα του 2012. Ήδη έχουμε μια σχετική ομάδα εργασίας για τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες και προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τις ε, βέλτιστες πρακτικές και θα προτείνουμε και κάποια μέτρα πολιτικών προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των κακών μαθητών σε ό,τι αφορά τι βασικέ δεξιότητε σε εθνικό επίπεδο. Επίση, ε, οι δράσει του προγράμματο Κομίνιου για το πρόγραμμα διαβίου κατάρτιση, μεταξύ των προτεραιοτήτων τη, περιλαμβάνει και την αύξηση των, του, ε, του ενδιαφέροντο για μαθηματικά και τεχνικέ επιστήμες και βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών. Η κυρία Μορκουνάιτε Μικουλένε για μισό λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την απάντηση. Μήπως έχετε κάποια στοιχεία για τις χώρες που έχουν τις ε, χειρότερες επιδόσεις στα σχολεία. Και για ποιους λόγους πιστεύετε ότι έχουμε τόσο κακές επιδόσεις σε ορισμένες χώρες. Υπάρχουν διαρθρωτικοί λόγοι, οικονομικοί και τι γνώμη έχετε για την στοιχειώδη εκπαίδευση. Γιατί η μελέτη του ΟΣΑ μιλά για τις μαθητικές επιδόσεις σε μέση και ανώτερη εκπαίδευση. Τι γνώμη έχετε για τη στοιχειώδη εκπαίδευση, κύριε Επίτροπε. Έχουμε μείνει πολύ πίσω, κύριε Επίτροπε. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, αν γίνεται. Μπορώ να σα δώσω λεπτομεριακά στοιχεία για τα κράτη-μέλη. Δεν έχουμε αναλύσει και συμπληρώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί δεν είναι δικό μα έργο να δούμε γιατί ορισμένα κράτη-μέλη έχουν χειρότερε επιδόσει από άλλα. Αυτό που κάνουμε πάντως στην ανάλυση μα είναι να προωθήσουμε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Και χαίρομαι ιδιαίτερω γιατί ορισμένε χώρε που ακολούθησαν τέτοιε καλέ πρακτικέ βελτίωσαν τη θέση τους από το 2006 και μετά σε ό,τι αφορά τους περισσότερες δείκτες του όσα. Σε ό,τι αφορά την ε, στοιχειώδη εκπαίδευση, τα δημοτικά δεν έχουμε αντίστοιχες μελέτες με αυτές της πίζα του όσα. Για τη βασική εκπαίδευση δεν υπάρχει τέτοια μελέτη για τα δημοτικά δυστυχώς. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ που ήσασταν ε, λακωνική, κυρία Επίτροπε. Θα περάσουμε τώρα σε ερωτήσεις προς την Επίτροπο Κρούς. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Κανονικά σε έξι λεπτά έπρεπε να έχουμε τελειώσει και έχουμε ερωτήσεις προς δύο επιτρόπους. Θα απαντήσουμε σε δύο ερωτήσεις ε, προς κάθε επίτροπο. Ερωτήσεις ε, Παπα-Νικολάου και Ελγόρτ προς την κυρία Κρούς. Κύριε Κρόλου, δυστυχώς τη δική σας δεν θα την ακούσουμε και ε, για τον κύριο Κάλλας θα απαντηθούν οι ερωτήσεις Πόσελ και Χίγγινς. Μόλις είναι έτοιμη η κυρία Κρούς, παρακαλώ να απαντήσει στην ερώτηση 19 του κυρίου Παπα-Νικολάου. Σας θέρμο παρακαλώ κύριε Επιτροπέ, κύριε Επιτροπέ και κύριοι συνάδελφοι, χρόνου φίδου, να είστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Mrs. Cruz, you have the Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη του 2020 και για την ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη, για 30 στόχοι για τη βασική ανάπτυξη για όλους τους Ευρωπαίους ε, μέχρι το 2030, έχει στόχο μέχρι το ε, να έχουν πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα όλοι οι Ευρωπαίοι από 30 MB ε, το δευτερόλεπτο και ε, μέχρι και 100 MB το δευτερόλεπτο. Γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει κίνδυνος πραγματικά στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που επικεντρώνεται η ευρυζωνικότητα μόνο σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και νησιά και αεροκατοικημένες είναι σε μειονεκτική θέση. Αυτό έχει να κάνει και με την εκπαίδευση και με την τεχνολογία ε, της πληροφορίας και τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι μόνο 67% των σχολείων έχουν ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο και υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη και πυκνοκατοικημένων και αεροκατοικημένων περιοχών. 73% ε, σε αντίθεση 60,6% οι αεροκατοικημένες. Για να μην ε, υπάρχουν προβλήματα, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει ένα πακέτο ε, ευρυζωνικότητας με εθνικές, πολιτικές και περιφερειακές για να φτάσουμε στους στόχους μας. Ε, αυτό θα μειώσει και το κόστος ε, της ε, γάλυψης ευρωζωνικής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμός και ε, να μειωθούν τα γραφειοκρατικά προσκόμματα. Έχει δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αυξηθούν οι επενδύσεις σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής έχουν προγραμματιστεί περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης της Οικονομίας ε, ε, έχει προβλέψει 360 εκατομμύρια ευρώ για την ευρυζωνική ε, ανάπτυξη της υπαίθρου. Στο πακέτο λοιπόν της ευρυζωνικότητας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι θα ενισχύσει και θα εξορθολογήσει τη χρηματοδότηση ε, μέχρι το 2014 και θα ε, διερευνήσει δυνατότητες προσέλκυσης ιδιωτικού κεφαλαίου ε, με ενίσχυση των πιστώσεων και των δανείων με ευρωπαϊκά κονδύλια και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αναμένεται λοιπόν πρόοδος κατά το 2011. Ένας άλλος πυλώνας της ψηφιακής ατζέντα, ε, κύριε Πρόεδρε, αναφέρεται στις ψηφιακές δεξιότητες. Για παράδειγμα, προτείνουμε ε, να μελετήσουμε ε, και να θεωρήσουμε τα στοιχεία αυτά προτεραιότητα για την κοινωνική χρηματοδότηση στην επόμενη προγραμματική περίοδο και να θεωρούμε τις ψηφιακές δεξιότητες συμπληρωματικές για μεγαλύτερη διαφάνεια στην παιδεία. Πώς γνωρίζετε η παιδεία είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην κοινωνία μας και συμφωνούμε ότι αν δεν υπάρξουν απαραίτητες επενδύσεις, ορισμένες περιοχές μπορεί να μείνουν πίσω τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 2006 και δείχνουν ότι μόλις 67% των σχολείων έχουν πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα και είναι πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πυκνοκατοικημένων και αραιοκατοικημένων περιοχών. Σε λίγο θα κάνουμε μια νέα μελέτη στα σχολεία και τα αποτελέσματα θα είναι έτοιμα τέλη του έτσι. Ο κύριος Παπα-Νικολάου, 32 σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε για την πολύ διεξοδική απάντησή σας. Συμπληρώνοντας, προσθέτω το εξής. Αναφέρουμε στην Ευρώπη για το 2020 στη στρατηγική μας ότι στόχος μας είναι μια ψηφιακή ενιαία αγορά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που σημαίνει ίσες ευκαιρίες για πρόσβαση, ίσες ευκαιρίες όμως και για ανάπτυξη. Εσείς οι ίδια κατά καιρούς σε ακροάσεις ε, στι αρμόδιε επιτροπέ, και το θυμάμαι και εγώ ίδιο στην επιτροπή Παιδεία και πολιτισμού μας αναφέρατε ότι για τα επόμενα πέντε χρόνια περίπου 500.000 νέες θέσει εργασία θα χρειαστούν στους τομείς αυτούς αν θυμάμαι καλά. Και ρωτώ συγκεκριμένα, λαμβάνουμε όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε η δημιουργία αυτών των θέσεων εργασία να κατανεμηθεί δίκαια χωρίς να αποκλεί τι γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές. Ευχαριστώ πολύ. Mr. President, the answer is yes. Κύριε Πρόεδρε, απάντηση είναι ναι. That's very good. Thank you very much indeed. Now we move to the question by Mr. Aylward on the 116 missing child. Στην ερώτηση του για την ε, γραμμή σχετικά με τα αγνοούμενα παιδιά της κυρίας Λάιαμ, γραμμή 11.6000. Κύριε Πρόεδρε, η εφαρμογή, ε, η εισαγωγή αυτής της τηλεφωνικής γραμμής απαιτεί περισσότερες προσπάθειες σε πολλά κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν έχουμε τους ε, Μιλάω κυρίως για το άρθρο 27 ε, της Οδηγίας περί Οικουμενικών Υπηρεσιών. Εκεί προβλέπεται τα κράτη-μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε αυτή την τηλεφωνική γραμμή και εκεί να αναφέρουν περιπτώσεις αγνοούμενων παιδιών. Ε, η Κομισιόν ελέγχει ε, και βοηθάει τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή αυτής της νέας διάταξης σε εθνικό δίκαιο, κάτι που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 25 Μαΐου του 2011. Στις 17 Νοεμβρίου του περασμένου έτους η Κομισιόν ενέκρινε αυτήν την τηλεφωνική γραμμή, ε, την 11.000 στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα γνώμενα παιδιά. Ο στόχος της ανακοίνωσης είναι να ε, ανανεωθεί η έκκληση της ε, Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη να λάβουν αυτό το θέμα ως προτεραιότητα και να διασφαλίσουν ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσφέρεται η ίδια ποιότητα υπηρεσιών, πρακτική υποστήριξη στα κράτη-μέλη και η ανακοίνωση προβάλλει τις βέλτιστες πρακτικές κρατών μελών ε, για ε, να ε, εφαρμοστεί αυτή η τηλεφωνική γραμμή, να λειτουργεί αυτή. Η ε, Κομισιόν προτείνει αυτές οι βέλτιτες πρακτικές να καταλήξουν σε ένα κοινό παρονομαστή που θα διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε οι γονείς και τα παιδιά να υπολογίζουν στην ίδια βοήθεια ανεξάρτητα που βρίσκονται. Ε, εδώ δεν πρόκειται μόνο για ηλεκτρονικά θέματα για τα οποία είμαι αρμόδια, ε, τα συντονίζει εξίσου και η συνάδελφος κυρία Ρέντινγκ την συμπληρωματική σας παρακαλώ κύριε Αλγούρ. Κατά το παρελθόν μιλήσατε ε, για το κόστος και για την έλλειψη πληροφοριών ως ε, εμπόδιο ε, να λειτουργήσει αυτή η τηλεφωνική γραμμή σε ορισμένα κρατημέλη. Τι θα κάνετε για να μην υπάρχουν πια αυτοί οι φραγμοί και θα μεριμνήσετε έτσι ώστε η γραμμή αυτή να υπάρχει σε όλα τα κρατημέλη και ποιε εναλλακτικέ λύσεις υπάρχουν σε κρατημέλη που δεν έχουν χρήματα να χρηματοδοτήσουν αυτή τη γραμμή έτσι ώστε να λειτουργεί και εκεί. Επίτροπος. Και βέβαια προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα για την ε, γραμμή αυτή. Πράγματι, ανέφερα παλαιότερα, το κόστος είναι ένα θέμα, αλλά δεν είναι η γραμμή ίδια αυτό είναι το ελάχιστο μέρος του προβλήματος. Το πρόβλημα είναι η συνέχεια και η συνέχεια έχει νόημα γιατί το να υπάρχει μόνο η γραμμή κύριε Πρόεδρε δεν είναι το μόνο θέμα στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Η συνέχεια παίζει ρόλο. Ελέγχουμε λοιπόν προσεκτικά και βοηθάμε τα κρατημέλη στην εφαρμογή και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ε, Αυτά πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με βάση τη σημερινή οικονομική κρίση είναι ακόμα πιο δύσκολο για ένα κράτος μέλος να αναζητήσει τρόπους χρηματοδότησης ε, της συνέχειας. Σε ορισμένους ε, οργανισμούς υπάρχει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αλλά δεν έχει ως στόχο να καλύψει το πλήρες κόστος απλά να βοηθήσει έτσι ώστε ε, να υλοποιηθεί αυτή η τηλεφωνική γραμμή και βεβαίως ε, πρέπει κανείς ε, να είναι παραγωγικός οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να είναι παραγωγικές να αναζητήσουν ε, πόρους, ε, εταιρική ευθύνη και δώρες, έτσι ώστε σε τελική ανάλυση να γίνει αυτό που θα θέλαμε όλοι μας τόσο πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θα περάσουμε τώρα σε ερωτήσεις προς τον Επίτροπο Κάλλας. Η πρώτη είναι του κυρίου Πόσελτ. Του σιδηροδρομικού άξονες των Άλπαιων αφορά και μόλις καθίσει ο Επίτροπος και είναι έτοιμος μπορεί να απαντήσει. Η επόμενη ερώτηση προς τον κύριο Κάλλας που θα είναι και η τελευταία του της απογευματινής συνόδου θα είναι του κυρίου Higgins για την αποστολή μηνυμάτων. Ο κύριος Κάλλας, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα των σιδηροδρομικών αξώνων των Άλπων είναι πολύ σημαντικό. Και δεν είναι και άσχημα τα πράγματα σε αυτή τη φάση. Παρά τις δυσκολίες που είχαμε από οικονομικής άποψης, ε, το, η σύραγγα του Μπρένερ φαίνεται ότι προχωρεί καλά. Επίσης είναι ύψιστη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέμα αυτό που πρόβλεψε ένα δισεκατομμύριο σχεδόν προπολογισμό για, για τη σύραγγα αυτή. Σε ό,τι αφορά την βασική σύραγγα του Μπρένερ, η Δικαιβερνητική Επιτροπή τη 19η Νοεμβρίου του 2010 παρουσία του Ευρωπαίου συντονιστού, Πατ Κόξ, ε, οδήγησε σε πολύ αισθητή πρόοδο και μάλιστα ε, συμφωνήθηκε το συνολικό κόστος 8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη βασική σύραγγα και μάλιστα η Αυστρία ε, ενέκρινε και βελτιστοποίησε το σχέδιο εργασιών που θα επιτρέψει την έναρξη των προπαρασκευαστικών εργασιών μέχρι το τέλη του 2011. Επίσης και η Ιταλική πλευρά συμφώνησε για τις εγγύησεις ό,τι αφορά το συνολικό κόστος. Υπάρχει λοιπόν πρόοδο και όσο ό,τι αφορά τι αναγκαίε γραμμέ πρόσβαση και στι δύο πλευρέ. Η Ιταλία ενέκρινε την έναρξη των εργασιών του Νοτίου Άξονα για το πρώτο τμήμα και μάλιστα πρόοδος έχει γίνει και από την Αυστρία για το πρώτο τμήμα που θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2013, και νωρίτερα. Σε ό,τι αφορά τι διασυνοριακέ διασυνδέσει ε, Αυστρία και Γερμανία. ο αρχικός στόχος του ολοκλήρωσης του έργου μέχρι το 2012 το αργότερο, Δυστυχώ δεν θα υλοποιηθεί. Σε ό,τι αφορά τη γερμανική πλευρά, τα έργα δεν θα, δεν θα αρχίσουν πριν το 2012 και θα διαρκέσουν τουλάχιστον μία τριετία. Πάντως η Γερμανία τον Νοέμβριο του 2010 δημοσίευσε την Εθνική Αξιολόγηση Επενδύσεων που περιλαμβάνει κάποιες θετικές εξελίξεις για τον βόρειο άξονα ε, Μονάχου και Αυστριακών Συνόρων. Θα ηλεκτροδοτηθεί το όλο τμήμα και το επόμενο βήμα θα είναι ένα μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Γερμανίας και Αυστρίας για τη διαχείριση των υποδομών αυτού του τμήματος και θα πρέπει μετά να ξεκινήσει και η κανονική διαδικασία προγραμματισμού. Σε ευχαριστώ. Ο κύριος Πόσελτ και μετά ο κύριος Χουντής. Ο κύριος Πόσελτ, πρώτος. Ευχαριστώ για την καλή σας απάντηση, κύριε Επίτροπε. Αλλά το δεύτερο σκέλος ερώτηση δεν μου το απαντήσατε. Για τη συνδρομική γραμμή Μόναχο Μίλντορ Φράι Λάσινγκ, που είναι τμήμα της γραμμής του ε, το Βουδαπέστη και είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, λόγω του βαβαρικού τριγώνου και ε, την αποσυμφόρηση προς τον Μπερένερ γιατί αν έρθει το τούνελ, η σύραγγα ε, του Μπρένερ ε, θα επιβαρυνθεί άλλος άξονας, γι' αυτό θα πρέπει να επεκταθεί η συνδρομική γραμμή Μόναχο Μίλντορ Φράιλασινγκ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο προτεραιότητας και φροντίστε στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές να δώσετε και πάνω χρηματοδότηση. Είναι διασυναριακό το έργο. Ο κύριος Χουντής παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εδώ μπροστά Κύριε Επίτροπε, ναι ωραία αυτά που γίνονται στις άλπεις αλλά στην ελλάδα λόγω του μνημονίου η ελληνική κυβέρνηση προχωράει σε περικοπές και διακοπές δρομολογίων που απομονώνουν την ελλάδα από το ευρωπαϊκό και το βαλκανικό σιδηροδρομικό δίκτυο επικαλούμενη και η κομισιόν και η ελλάδα ότι ο οργανισμός σιδηροδρόμων της ελλάδας έχει μεγάλο χρέος. σας ερωτώ λοιπόν πώς κρίνετε αυτές τις εξελίξεις τις περικοπές δηλαδή των σιδηροδρομικών δρομολογίων και δεύτερο αν στο χρέος του οργανισμού των σιδηροδρόμων της ελλάδας θεωρούνται ότι είναι και τα χρήματα για να συγχρηματοδοτούμε τα έργα υποδομή μαζί με την ευρωπαϊκή ένωση. ευχαριστώ πολύ. Ε, νομίζω ότι η Ελλάδα προχώρησε πολύ, έφτασε πολύ πιο κοντά στις Άλπεις από ό,τι νόμιζα εγώ. Για την Ελλάδα. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Και δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση για τα προβλήματα αυτά. Σε ό,τι αφορά τη γραμμή μονάχου Μίλτορφ Φράιλασινγκ Σάλσμπουργκ, το σχέδιο προτεραιότητας υπαριθμό 17, καλά πάει. Άρχισαν ήδη οι προεργασίες το 2007 και μερικά έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Το νέο, νέος άξονας διπλής κυκλοφορίας έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Μίλντορφ και θα ολοκληρωθεί όσον Καλύπτεται από το γερμανικό σχέδιο ανάκαμψης με 11,7 εκατομμύρια. Ανα... Εξελίσσεται το σχέδιο αυτό λοιπόν της σιδηροδρομικής γραμμής. Δεν δημιουργεί προβλήματα, ειδικά αυτή η γραμμή. Προ το παρόν τουλάχιστον. Καλώ και πέραμε στην τελευταία ερώτηση τη βραδιά, του κυρίου Χίγγινς, ε, την αποστολή ανταλλαγή μηνυμάτων στο κινητό κατά την ώρα τη οδήγηση. Κύριε Κάλλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Βουλευτά και κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη ε, του κυρίου Χίγγινς ότι η αποστολή μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο την ώρα τη οδήγηση. Ε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη όπως γνωρίζετε το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε μία έκθεση ε, για τη ε, χρησιμοποίηση των κινητών την ώρα της οδήγησης και έχει δημοσιευθεί και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. Δεν υπάρχουν στατιστικές για τον αριθμό των ε, ατυχημάτων που οφείλονται ακριβώς αυτό. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν νομοθεσία που απαγορεύει τη χρήση του κινητού και στο διαδίκτυο και την αποστολή μηνυμάτων και τα πάντα. Ένας οδηγός θα πρέπει να είναι πλήρως συγκεντρωμένος στη οδήγηση την ώρα που οδηγεί και να μην αποσπάται η προσοχή του από άλλες δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, προτίστε να επιβάλλει και ένα, άλλο στρώμα ευρωπαϊκής νομοθεσίας πάνω από τα εθνικά στρώματα για να απαγορεύεται το διαδίκτυο, το browsing, το, η αποστολή μηνυμάτων ε, γραπτών από τα κινητά κτλ. Ελπίζουμε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό ε, αρμοδίως. Ο κύριος Χίγκινς και μετά ο κύριος ε, Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απογοητεύομαι από αυτά που μου απαντάει ο Επίτροπος κύριος Κάλλας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργάζονται τα διάφορα κράτη-μέλη και να προσπαθούν να καταλήγουν σε κάποια συμφωνία. Θα πρέπει να μειώσουμε τα θανατηφόρα τροχέα και τα σοβαρά τροχέα που προκαλούν πολλούς τραυματίες. Οι νέες τεχνολογίες ε, ενοχλούν ε, και παρεμποδίζουν την οδήγηση. Οι κανόνες στα κράτη-μέλη διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Απογοητεύομαι πάρα πολύ από αυτό που μας λέτε, ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας απαντήσει περισσότερο. Ευχαριστώ. Κύριος ε, Κέλλη. Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Χίγγινς που έθεσε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Συμμερίζομαι και εγώ την ανησυχία του και την έλλειψη, για την έλλειψη ενθουσιασμού από πλευρά Επιτρόπου για τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να επιβληθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορείτε τουλάχιστον να προσπαθείτε να ενθαρρύνετε περισσότερο τα κράτη-μέλη να έχουν τους ίδιους κανόνες και την ίδια νομοθεσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιβάλλεται η νομοθεσία και να εφαρμόζεται προς όφελο όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος. Α, συγγνώμη. Η κυρία Γιάλα. Πάρα πολύ σύντομα. 30 δεύτερα παρακαλώ. Ναι, το μόνο που θέλω να πω είναι να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι είμαι εισηγήτρια ακριβώς ε, του θέματος για τις διασυνοριακές ε, ενώσεις τους άξονες για να μπορέσει ε, για τις παραβάσεις συγγνώμη, τις διασυνοριακές ε, που είναι και αυτό το θέμα ε, της χρήσης των κινητών αλλά δυστυχώς άλλαξε η νομική βάση το Συμβούλιο και ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο ούτε η Ιρλανδία ε, συμμετέχουν γιατί έχουν opt-in out. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ίσως στο Κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και ελπίζω στη συζήτηση με τις χώρες αυτές να προχωρήσει. Ε, φαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να μπει στο σύστημα, αλλά δεν έχουν προχωρήσει πολύ τα πράγματα. Ευχαριστώ. Κύριε Κάλλας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ το πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια και εφαρμογή του ήταν πολύ μεγάλη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πραγματικά ε, οδήγησε σε τεράστια πρόοδο, τεράστια ουσιαστικότατη μείωση των ε, δυστυχημάτων έχουμε στην Ευρώπη. Και στη χώρα μου, στι αρχέ του 90 πρέπει να σας πω ότι είχαμε 400 θύματα το χρόνο. Πέρυσι ήταν μόλι 78 τα θύματα των τροχαίων. Και ε, μειώθηκε ε, ο αριθμός αυτός ενώ δεκαπλασιάστηκαν και πλέον τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και ευχαριστώ την κυρία Γιάλα που επιθυμίζει τη διασυνοριακή εφαρμογή και η συνέχεια που δίνεται στις παραβάσεις είναι πολύ σημαντικό αυτό για να αυξηθεί η οδική ασφάλεια. Η σχετική απόφαση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Λήφθη το Δεκέμβριο και είμαστε στο στάδιο της εφαρμογής της. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι η αύξηση των νομοθετημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μια πανάκια. Δεν είναι απάντηση σε όλα ότι ό,τι πρόβλημα και να έχουμε βάλει μια ευρωπαϊκή ε, νομοθεσία. Γιατί θα καταντήσουμε να έχουμε υπερβολική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ήδη δεχόμαστε κριτικές γι' αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα των κρατών μελών και τη κοινή γνώμη και ανησυχεί ο κόσμος ε, γενικά για αυτά τα θέματα. Και μπορούν να αντιμετωπιστούν διασυνοριακά και να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός χώρος οδικής ασφάλειας, έτσι ώστε οι παραβάσεις να διαπιστώνονται διασυνοριακά και τα πρόστιμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους διερμηνείς και το προσωπικό. Διακόπτεται η συνεδρίαση και θα επαναληφθεί στι 9.